Καλημέρα σα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ε, ξεκινάμε σιγά σιγά. Έχουν φτάσει περισσότεροι συνάδελφοι, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε. Σημείο πρώτο. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε καμία παρατήρηση. Όχι, οπότε θεωρώ ότι εγκρίνεται. Ε, μεταδίδεται και στο διαδίκτυο η σημερινή μας συνεδρίαση και έχουμε διερμηνία σε 16 γλώσσες. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 22ης και 23ης Ιανουαρίου. τόσο λίγο θα ψηφίσουμε και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προώθηση των Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών και την ε, παρότριση του κλάδου να παράγει περισσότερες πρωτεΐνες καλλιεργώντας πρωτεϊνούχα και ψυχανθή είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα των πρωτεϊνούχων και ψυχανθών φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα των ζωοτροφών, τα ψυχανθή και τα πρωτεϊνούχα προϊόντα. Οπότε ε, είναι η βάση για, για έναν από τους βασικούς ε, τομείς της ευρωπαϊκής παραγωγής, της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας. Είμαστε στην αρχή και όχι στο τέλος μιας ε, μακροχρόνιας διαδικασίας, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ε, πρόθεση μέχρι το τέλη του 2018 να υποβάλει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τις Πρωτεΐνες ε, και περαιτέρω πρωτοβουλίες που θα εγκαινιαστούν από το 2019 και μετά. Οπότε η δική μας έκθεση πρωτοβουλίας στόχο έχει την της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλάβει πιο εκτεταμένες δράσεις και πρωτοβουλίες υπέρ της καλλιέργειας πρωτεϊνούχων και ψυχανθών. Και μάλιστα η Βουλγαρική Προεδρία σκοπεύει να περιλάβει ε, το θέμα αυτό στο επόμενο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε να λάβει υπόψη και τη δική μας έκθεση πρωτοβουλίας στις προτάσεις της. Βέβαια, πιο αρμόδιος για να επεκταθεί σε λεπτομέρειες για το θέμα αυτό είναι ο συντάκτης της έκθεσης, ο κύριος Ζων Πολ Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα ουσιώδη τα καλύψατε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας. Ε, δεν θα επιμείνω περισσότερο σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους ε, συνεταιρισμούς, γεωρικούς συνεταιρισμούς, ε, τους κτηνοτρόφους, τους επιστήμονες που συνέβαλαν στην διαμόρφωση της έκθεσης, αλλά και τους και ηγητές που με τις τροπολογίες τους εμπλούτησαν την έκθεση και μας επέτρεψαν, ελπίζω, να βρούμε μια καλή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων θέσεων. Και ευχαριστώ και τους συνεργάτες μας για τη βοήθειά τους. Πιστεύω ότι σήμερα αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας προτείνει σημαντικές ιδέες για το πρωτεϊνικό ζήτημα στην Ευρώπη. Και σας καλώ να περάσουμε στην ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τενανό, και να καλωσορίσω και πάλι τους συναδέλφους και τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας προτείνω να περάσουμε στην ψηφοφορία. Πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τροπολογία 1 του κυρίου Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1, και πιστεύω ότι έχει απορριφθεί. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Της κυρίας Πετήρ και του κυρίου Ντες. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 281. Ποιος είναι υπέρ της 281. Κατά. Απορρίπτεται. 282. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 127. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν και μάλλον απορρίπτεται. Τέλος ψηφοφορίας. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, συγγνώμη λέει ο Συμβαστική τροπολογία 3 πρώτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Κάποιο ζητά έλεγχο της προηγούμενης τροπολογίας. Καλώς, οπότε ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 33, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Αν και ήταν οριακή διαφορά, οπότε εύλογη η πρόταση για εξακρίβωση του αποτελέσματος. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 5 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Περνάμε στην παράγραφο 4 και την τροπολογία 147. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 148. σαράντα οκτώ. Α, όχι. Εκατόν Πάμε στην 152. Ποιος είναι υπέρ. Όχι, προηγείται ηλεκτρονικός έλεγχος της τροπολογίας 147. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην 152 Κατά. Όχι, μάλλον διόρθωση. Επειδή η 147 έχει απορριφθεί, πρέπει να ψηφίσουμε και τις ακόλουθες. Οπότε περνάμε στην 148. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 148. Τέλος. Απορρίπτεται. 149. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 149. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Οπότε τώρα περνάμε στην 152. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία γιατί είναι συμβαστική τροπολογία 6. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται. 164 του κυρίου Χόισλινγκ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 164. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στη συμβαστική τροπολογία 6 ή μάλλον 7 διορθώνει ο πρόεδρος, 7 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 172. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 175. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 176 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 177. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 177 της ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 178. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 181. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 181. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 182. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 183 υπέρ. πάμε κατευθείαν στη συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 193. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 194 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Διακόσια πέντε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται μάλλον να το ελέγξουμε καλό κακού. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 10, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 202. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 212. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 212. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. απορρίπτεται. Πάμε στην 215. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 216. Ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται, αλλά θα το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. απορρίπτεται. 217. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 12. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Μάλιστα. 2.24 ε, της κυρίας Νταντζίλα που είναι, έγινε και πρωθυπουργός στο μεταξύ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στη 233 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 235. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 247. Συγγνώμη, μια διόρθωση. Πάμε στην τροπολογία 32 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τώρα συμβαστική τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 247. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ελεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 248. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 249 υπέρ κατά απορρίπτεται. 250 υπέρ κατά απορρίπτεται. 252 υπέρ κατά απορρίπτεται. 253 υπέρ εγκρίνεται. 255 υπέρ εγκρίνεται. 256 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 34 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ εγκρίνεται. 259 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 285. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 29 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Ελάχιστα σηκώνατε το χέρι, γι' αυτό έπρεπε να ελέγξουμε. 2,89. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 336. Ποιος είναι υπέρ. Α, όχι. Εγκρίνεται, εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. Πάμε στην 18α. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Και τώρα συμβαστική τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 297. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 298 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 300 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 20. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 309. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 309. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 312. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 312. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 326. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 326 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 337. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 204. Τον Καπούτο και Ντενανό. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Οπότε δεν πάμε στην 29, αλλά κατευθείαν στη συμβαστική τροπολογία 22. Άρχεται ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 22. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 του κυρίου Χόισλινγκ υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. του κυρίου Χόισλινγκ τροπολογία. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Εγκρίνεται. 22α. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί μερικοί δεν ψηφίζουν. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22α. α. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 23. Υπέρ. Άρχεται ψηφοφορία, συγγνώμη. Τέλος. Εγκρίνεται. εδώ περάμε στην τροπολογία 28. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 28. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 28. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 24. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 25. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται και πάμε στη στην συμβαστική τροπολογία 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Όχι. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 28. Άρχεται ψηφοφορία. Ή θέλετε έλεγχο προηγουμένως για την 54. Καλώς επαναφορά στην 54 και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για έλεγχο. Τροπολογία 54, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Όντως απορρίπτεται. Συμβεστική τροπολογία 28. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 84. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 86. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 32. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 88. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 110. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 92. Ποιος είναι υπέρ. Ε, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 33. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 99. 99. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην 106 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος 106 κατά απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται και αυτό. Πάμε στην 107. Ποιο είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά απορρίπτεται. 109 υπέρ εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά απορρίπτεται. 114. 115. Λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περιλαμβάνεται στην συμβαστική τροπολογία 27. 114. Αυτό μου εξηγεί η γραμματεία. Οπότε Λυπάμαι που δεν αναφέρεται στο κατάλογο ψηφοφορία ε, αυτή η υπόμνηση. Υπερψηφίσαμε την 27, αλλά δεν ψηφίζουμε τον 114. Και τώρα περνάμε στο σύνολο της ε, έκθεσης με τις τροπολογίες. Ή μάλλον πρώτα την 115. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης ε, όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ντενανό. Έχετε το λόγο αν θέλετε. Α, χειροκροτήματα εν είδη ευχαριστίων. Ο κύριος Ντενανό. Ή μήπω δεν θέλει. Ναι, ήθελα απλά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και ελπίζω ότι και στην Ολομέλεια η ψηφοφορία θα είναι ανάλογη και αυτό θα βοηθήσει και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιών και ότι το Κοινοβούλιο θα κάνει τη φωνή να ακουστεί για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Ντενανό. Ευχαριστούμε και τους και και τους συνεργάτες και πάλι συγχαρητήρια στον εισηγητή. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε με το σημείο 5. Ένα λεπτό διάλειμμα.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 Przechodzimy do punktu kolejnego. Πάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 5 και καλωσορίζω τους συναδέλφους, τους καλεσμένους μας μάλλον από την Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας παρουσιάσουν την έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των διεθνών δραστηριοτήτων που αφορούν την καλή διαβίωση και καλή μεταχείριση των ζώων στην ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παραγωγών ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας, οι συντονιστές αποφάσισαν να ζητήσουν από την Επιτροπή να μας παρουσιάσει την πρόσφατη έκθεσή της με αυτό το θέμα, δηλαδή τον αντίκτυπο των διεθνών δραστηριοτήτων που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων στην ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων ακτινοτρόφων. Και μάλιστα σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Ε, είναι προφανής η σημασία του θέματος αυτού για τους Ευρωπαίους παραγωγούς κρέατος, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέκαθεν ε, στην πρώτη γραμμή, ευαισθητοποιώντας παγκοσμίω για την ανάγκη καλής μεταχείρισης των ζώων και έχοντας ένα αξιόπιστο κανονιστικό μοντέλο για το θέμα αυτό. Καλό όμως ε, θα ήταν το μοντέλο μας αυτό το νομοθετικό να επεκταθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε οι καλές μας προδιαγραφές και πρακτικές να εφαρμόζονται και παγκοσμίω. Και καλό θα ήταν ε, και η κοινή γνώμη να ασκήσει πίεση υπέρ της ε, εξάπλωσης αυτών των προδιαγραφών. Οπότε καλό είναι να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση και να θαρρύνουμε τους ε, εμπορικούς μας εταίρους παγκοσμίω υπέρ της καλής μεταχείρισης των ζώων. Και μάλιστα έχουμε πολλές δραστηριότητες και εντός και εκτός της Ένωσης ε, με δοκινοτικού και εξοκινοτικούς παραγωγούς για τα θέματα αυτά. Ένας εκπρόσωπος Γενικής Διεύθυνσης ε, Υγείας ε, θα μας παρουσιάσει την πρόσφατη έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Εσκριβάνο θα μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση εδώ για να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση. Το 2012 η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προστασία και την Ευημερία των Ζών ε, περιλάμβανε 12 δράσεις, μέχρι των οποίων και αυτή η έκθεση. Η έκθεση αυτή βασίζεται σε μια προπαρασκευαστική μελέτη για τον αντίκτυπο ε, της ευμαρίας των ζώων και, των σχετικών διεθνών δραστηριοτήτων. Η προώθηση της ευημερίας των ζώων είναι ε, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θέλουμε να έχουμε ψηλά πρότυπα τα οποία θα αποτυπώνουν τις ευρωπαϊκές αρχές και το ευρωπαϊκό μοντέλο. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή για να προωθήσει ένα μοντέλο το οποίο αποφασίζεται επιστημονικά στοιχεία και το οποίο πλέον ασπάζονται πολλέ άλλε χώρε. Έχουμε, έχουμε όμω περιορισμένε αρμοδιότητε σε ό,τι αφορά τι μη ευρωπαϊκέ χώρε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε και να έχουμε ε, ισχυρέ ε, σχέσει με διεθνού οργανισμού, οργανισμούς που έχουν ε, εντολή προ την κατεύθυνση αυτή και των οποίων οι δράσει είναι συμπληρωματικέ. Βλέπετε εδώ ποιες ε, δράσεις χρησιμοποιούμε, διασκέψεις, ε, δημιουργία δυνατοτήτων, ε, κατάρτιση, θα επανέλθουμε από αυτού. Η έκθεση επικεντρώνεται στις βασικές δραστηριότητε που διεκπεραιώνει η Κομισιόν με την υποστήριξη των κρατών μελών. Ο στόχος είναι να εξετάσουμε το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την προώθηση των προτύπων της ευημερίας των ζώων παγκοσμίω και να αναλύσουμε την συνεισφορά αυτών των δραστηριοτήτων έτσι ώστε να υπάρξει ε, ένα δίκαιο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ευρωπαίων και μη Ευρωπαίων ε, κτηνοτρόφων. Λαμβάνουν χώρα και σε πολυμερές και σε διμερές επίπεδο οι δραστηριότητες μας. Σε πολυμερές επίπεδο θέλουμε να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη διεθνών προτύπων από την Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων, τον OIE. Από κοινού με τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρουν στην διαδικασία θέσπιση προτύπων για να εξασφαλίσουμε ότι οι αρχέ μα θα ε, γίνονται σεβαστέ στο μέτρο του δυνατού. Τεχνική πραγματογνωμοσύνη, ε, συμμετοχή στι διάφορε ομάδε. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση και υποστήριξη τη εφαρμογή των προτύπων OIE σε χώρες εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, έχουμε υποστηρίξει σε τεχνικό επίπεδο δραστηριότητες του ΟΑΗ, e τις έχουμε χρηματοδοτήσει, έχουμε αυξήσει τον προπολογισμό μας ε, που αφιερώνεται σε ζητήματα ευημερίας των ζώων στον ΟΑΗ. E. Αυτά τα πρότυπα του ΟΑΗ e είναι η βάση για μια κοινή κατανόηση με τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γενικότερα προωθούμε τα πρότυπά μας μέσω της δραστηριοτήτων δημιουργίας δυνατοτήτων capacity building, ε, το TIEX, ε, η FAO, η FAO, ο ΦΑΟ μας βοηθάει στο έργο αυτό. Πέρα από τα, τη θέσπιση διεθνών προτύπων, που είναι βασική δραστηριότητα και πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 14 πρότυπα για την ευημερία των ζώων, η Κομισιόν παρακολουθεί ε, την εφαρμογή των περιφερειακών στρατηγικών του ΟΑΗ και βεβαίω υποστηρίζει οικονομικά αυτέ τι στρατηγικέ όχι μόνο τι παρακολουθεί και τι προωθεί. Έχουμε μια στρατηγική ε, σφαιρική παγκόσμια για την ευημερία των ζώων που τυχάνει υποστήριξη από τους διεθνείς οργανισμούς, δημιουργεί ε, εταιρικέ σχέσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι βασικός ε, δωρητή των ΟΑΗ και πολλέ δραστηριότητε έχουν χρηματοδοτηθεί μεταξύ των οποίων η πλατφόρμα για την ευμερία των ζώων στην Ευρώπη. Αυτή η πλατφόρμα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Ευρώπης, γιατί καλύπτει ε, περιοχές όπου εμείς ε, δεν έχουμε αρμοδιότητα, όπως το θέμα των αδέσποτων σκυλιών, παραδείγματο χάρη. Επίσης έχουμε κοινέ δράσεις με τον ΦΑΟ, όπου προσπαθούμε να προωθήσουμε την ευμερία των ζώων ως δημόσιο αγαθό, σε διμερές επίπεδο, οι στόχοι μας είναι πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε ότι η εφημερία των ζώων θα περιλαμβάνεται σε όλες ε, τις ε, εμπορικές συμφωνίες που είναι υποδιαπραγμάτευση με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ε, και η εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί στα διάφορα φόρα συνεργασίας, με βάση διάφορου διακανονισμού. Βλέπετε εδώ τον κατάλογο των χωρών ε, με τι οποίε υπάρχουν τέτοιε συμφωνίε. Ε, η βασική στόχη σε διμερέ επίπεδο είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να υπάρχει, η ευαισθητοποίηση και να υπάρχει μια κοινή ε, αντίληψη για τα ζητήματα ευημερία των ζώων, να μοιραστούμε τι τεχνικέ μα γνώσει γνώσεις που μας ζητούν όλο και περισσότερο οι μη ευρωπαϊκές χώρες, να υποστηρίξουμε και να αναπτύξουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας περί των ζώων, εφαρμόζοντα τα πρότυπα ε, της, ε, του ΟΑΗ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συζητούμε και συζητήσεις, να συζητούμε μάλλον και ζητήματα που έχουν αντίκτυπο στο εμπόριο και που σχετίζονται με την ευμερία των ζώων. Επίσης έχουμε έντονη δραστηριότητα σε επίπεδο έρευνας, ε, τεχνικής συνδρομής και δημιουργίας δυνατοτήτων. Βλέπετε εδώ τις βασικές δραστηριότητες για την περίοδο 2004-2015. Νομίζω ότι μπορείτε εδώ να εκτιμήσετε την προσπάθεια που έχουμε καταβάλει έτσι ώστε να προωθήσουμε την ευμερία των ζώων παγκοσμίω. Ένα άλλο σημαντικό μέρος αυτής της μελέτης έχει να κάνει με τον αντίκτυπο για την ανταγωνιστικότητα. Όπως είπα στην αρχή της παρέμβασής μου, αυτή η έκθεση βασίζεται σε μια μελέτη. Και το σκέλος που αφορά την ανταγωνιστικότητα ε, πρέπει να πω εδώ ότι είχαμε ένα περιορισμένο αριθμό απαντήσεων για να αναλύσουμε το αποτέλεσμα, οπότε ε, επειδή δεν είχαμε τόσες απαντήσεις, δυστυχώς ε, τα αποτελέσματα αυτά ε, θα πρέπει να ληφθούν, να ληφθεί υπόψη αυτή η έλλειψη επιπτώσει απαντήσεων για να τα εκτιμήσουμε. Εξετάζουμε εδώ ποιοι τομεί επηρεάζονται από τα ζητήματα ευημερία των ζώων και ποιο είναι ο αντίκτυπο τη συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά σε τέσσερις ε, διαστάσεις κλειδιά της ανταγωνιστικότητας. Πρώτα, το θέμα της παραγωγικότητας και του κόστους ανταγωνιστικότητας. Εδώ υπάρχει διαφορά στην αντίληψη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, και κτηνοτρόφων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους Ευρωπαίους κτηνοτρόφους υπάρχει η αντίληψη ότι δημιουργείται ένα μειονέκτημα, ενώ για τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει το αντίθετο. Υπάρχει βεβαίως και το θέμα του θετικού αντικτύπου της συμμόρφωσης. Ε, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά το κόστος ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει να κάνει κυρίως το κόστος της ζωοτροφής και το εργασιακό κόστος και δεν έχει τόσο μεγάλη σχέση εδώ ε, το, τα πρότυπα, δεν, έχουν τόσο, δεν επηρεάζουν τόσο τα πρότυπα ε, ευημερίας των ζώων. Δηλαδή οι άλλοι δύο παράγοντες ε, είναι πολύ πιο σημαντικοί. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά τώρα, ε, η μελέτη δείχνει ότι η συμμόρφωση με την νομοθεσία περί ευημερίας των ζώων έχει θετικό αντίκτυπο για την πρόσβαση σε νέες αγορές και για τους ξενοτρόφους εντό και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ε, και για την πρόσβαση σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για κτηνοτρόφους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενδιαφέρον το αποτέλεσμα αυτό νομίζω. Σε ό,τι αφορά τώρα τις τρευλώσεις, τις εμπορικές, τρευλώσεις στην αγορά, δεν έχουν εμφανιστεί τέτοια φαινόμενα από τη μελέτη και σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα καινοτομία δεν μπορέσαμε ε, να ποσοτικοποιήσουμε εδώ, να εκτιμήσουμε την οικονομική σημασία ε, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα τα οποία είναι φιλικά προς τα ζώα, ας πούμε, ή που ε, σέβονται κάποιους κανόνες σχετικά με τα μεταχείριση των ζώων. Αυτό στα συμπεράσματα τώρα, ε, πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ε, προσέγγιση συνεργασίας ε, σε ό,τι αφορά την προώθηση των ε, ε, τη ευημερία των ζώων στη διεθνή σκηνή. Οι διεθνεί δραστηριότητέ μα ε, είναι μακροπρόθεσμη επένδυση, βασίζεται σε τρία στάδια. Πρώτα απ' όλα ευαισθητοποίηση, στη συνέχεια δημιουργία δυνατοτήτων και τέλο χρηματοδότηση. Όπω γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει σημαντικού πόρου για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη-μέλη, έχει παίξει έναν ε, πολύ σημαντικό, ε, αποφασιστικό ρόλο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης παγκοσμίω ό,τι αφορά ε, την ευημερία των ζώων με σημαντικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεσμεύεται ε, για ένα διεθνές εμπόριο που βασίζεται σε συγκεκριμένες αξίες όπως προβλέπεται και στην στρατηγική εμπόριο για όλους. Τα πρότυπα αυτά τα ευρωπαϊκά για την ευημερία των ζώων ήταν πηγή έμπνευση για πολλές εθελοντικές πρωτοβουλίες του κλάδου. Έχουμε καταφέρει να συμπεριλάβουμε την ευημερία των ζώων στον διάλογο με πολλές τρίτες χώρες και σε πολυμερές επίπεδο δραστηριότητες στα πλαίσια διεθνών οργανισμών ε, έχουν σίγουρα προωθήσει το μοντέλο περιευμερίας των ζώων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση για την προώθηση και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του OIE. Είναι ε, βασικό μέλο ε, που συνεισφέρει ε, για τη δημιουργία των προτύπων OIE. Επίσης έχουν παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τα πρότυπα αυτά εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και στα σφαγεία αλλά και κατά τις μεταφορές. Σε ό,τι αφορά τώρα τη, διεθνή, τη διμερή συνεργασία, έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες μεταχείρισης των ζώων σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει διευκολύνει και την εφαρμογή των απαιτήσεων περί εισαγωγών ε, σε ό,τι αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή. Τέλος, οι δραστηριότητες έρευνας, κατάρτισης και δημιουργίας δυνατοτήτων έχουν αγγίξει χιλιάδες επαγγελματίε, έχουν αυξήσει τις δεξιότητες, τις γνώσεις των ανθρώπων αυτών για το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων και έχουμε υποστηρίξει την εφαρμογή πολιτικών που είναι προς όφελος των ίδιων των χωρών αυτών. Τα πρότυπα Καλή μεταχείριση των ζώων έχουν περιορισμένο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παραγωγών στην παγκόσμια αγορά. Το συνολικό κόστος συμμόρφωσης με τα πρότυπα καλή μεταχείριση των ζώων παραμένει πολύ χαμηλό όταν εξετάζουμε τα, τους άλλους παράγοντες κόστους παραγωγής που επηρεάζουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και ε, τους, ε, τις διάφορες ε, τάσεις στην, στο παγκόσμιο εμπόριο. Επίσης η παγκόσμια προώθηση των, προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι την καλή μεταχείριση των ζώων συνεισφέρει στο μακροπρόθεσμο στόχο για να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των ζώων παγκοσμίω και να, μειωθεί, να μειωθούν οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Είναι μια ευκαιρία να προωθηθούν περαιτέρω αυτά τα πρότυπα. Ελπίζω αυτή η παρουσίαση να ήταν ενδιαφέρουσα για σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε όποια ερωτήματα. Σας ευχαριστούμε κύριε Σκριβάνο. Φαντάζομαι θα υπάρχουν απορίες κυρία Ράζ Γκαρσία πρώτα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ένα μισή λεπτό ο καθένας πάνω κάτω. Ευχαριστώ. Εγώ δεν συμφωνώ και πολύ με την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι η ανάλυση που κάνατε παρά είναι απλοϊκή. Γιατί δεν υπάρχει συνάφεια μεταξύ των δικών σας λεγόμενων και των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τους παραγωγούς. Εσείς μας είπατε ότι το κόστος καλής μεταχείρισης των ζώων και της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής ε, παγκοσμίω ε, είναι το μικρότερο τμήμα. Αυτό όμως παρά είναι απλοϊκό και υπεραπλουστευμένο, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το κόστος της καλής μεταχείρισης των ζώων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κόστος άλλων προδιαγραφών, όπως της επιστηστικής ασφάλειας ή του σεβασμού του περιβάλλοντος ε, που εφαρμόζουμε επίσης. Και από αυτή την άποψη δεν είμαστε και τόσο ανταγωνιστικοί, όλο και χάνουμε σε ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι ηλιοφαϊνότερο πια. Έχουμε προβλήματα με την πρόθεση των παραγωγών μας, ε, ε, ιδιαίτερα στην ανταγωνιστικότητα με τρίτες χώρες, ε, τις οποίες εισάγουμε και όλα. Εμείς έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες που δεν μιλούν μόνο για τις εκμεταλλεύσεις, αλλά και για τη μεταφορά των ζώων, μιλούν για τη σφαγή των ζώων. Και επίσης έχουμε ειδικούς, ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένους για παράδειγμα τις οτόκες όρνηθες, ή καλή μεταχείριση των ε, χείρων, ιδιαίτερα προς αναπαραγωγή. Το θέμα δεν είναι να πολλαπλασιάζουμε τους κανόνες μας και να θεσπίζουμε συνεχώς καινούργιους. Το θέμα είναι ότι οι υπάρχοντες κανόνες δεν εφαρμόζονται ομοιόμορφα ή στον ίδιο βαθμό σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης. Δεν χρειαζόμαστε νέους κανόνες, αλλά καλή εφαρμογή των ισχυόντων. Και επίσης, ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες, θα πρέπει να μεριμνήσουμε και να ε, βεβαιωθούμε ότι οι τρίτες χώρες που εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές και τους ίδιους κανόνες αυτό θα πει αμοιβαιότητα. Γιατί εμείς δεν έχουμε ε, τρόπους να εξακριβώσουμε την ε, ισχύ της αμοιβαιότητας. Αντί να θεσπίζετε νέους κανόνες, καλό θα ήταν να προβλέψετε μηχανισμούς ώστε να ελέγξουμε κατά πόσο οι τρίτες χώρες προσαρμόζουν τον τρόπο παραγωγής στις δικές μας αυστηρότερες προδιαγραφές και κανόνες και διατάξεις. Ευχαριστώ. Παρακαλώ 1,5 λεπτό καθένας, όχι παραπάνω. Κυρία Σλάιερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε η πρώτη συνάδελφος. Είμαι υπέρ βεβαίως της καλής μεταχείρισης των ζώων Καθώς προέρχομαι από τις ε, κάτω χώρες με πολύ μεγάλη παραγωγή, βέβαια ε, ανταγωνισμός ε, σωστός δεν υπάρχει πάντα, για τη μεταφορά έχουμε πάντα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις βεβαίως. Αλλά, και επισημαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλο ρόλο ο τομέα των μεταφορών, δεν γίνονται σεβαστοί πάντα οι κανόνες και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προβληθεί ο ρόλος των μεταφορέων. Εάν ωστόσο επιβάλλουμε επιπλέον απαιτήσει, θα αλλοιωθούν οι συνθήκες παραγωγής κρέατος που παράγεται σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Γιατί και εδώ επισημαίνω το έλλειμμα, ε, πρέπει να γίνει λόγος στη συμπεριφορά του παραγωγού. Πρέπει και αυτό να το συζητήσουμε αν θέλουμε να δείξουμε ποια είναι η θετική συμβολή της δικής μας παραγωγής. Κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Έχω ένα ερώτημα. Ενδιαφέρουσα η έκθεση. Ε, λέτε στα συμπεράσματα ότι αυτά τα πρότυπα ε, έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα. Πώς αξιολογήσατε τον αντίκτυπο σε ό,τι αφορά του ευρωπαϊκού παραγωγού. Πώ έγινε η αξιολόγηση, Είναι απλώ ε, μία έρευνα με περιορισμένα στοιχεία, υπάρχουν κάποιε άλλε παράμετροι. Δεύτερον, ποιο κριτήριο ε, ισχύει σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη στι διεθνεί εμπορικέ συμφωνίε, διότι από ό,τι μαθαίνουμε Κάπου έχουμε πρόοδο, κάπου άλλο όμως πάλι όχι. Στις με την Αφρική δεν γίνεται σχετική αναφορά με την, με την Νότιο Αφρική ούτε με τη Βόρεια Αφρική. Δεν φαίνεται να υπάρχει εκεί κάποια αναφορά σε αυτά τα πρότυπα. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι αυτά τα κριτήρια συμπερίληψης και γιατί ε, με κάποιες χώρες υπάρχει ε, συμπερίληψη και με κάποιες άλλες όχι. Σε ό,τι αφορά τώρα το συμπερίληψη του προτύπου στους διεθνείς οργανισμούς αυτό είναι θετικό ε, σε ό,τι αφορά τον ΟΑΗ ε και τον ΦΑΟ είπατε αναφερθήκατε κυρίως στη σφαγή ε, και στη, μεταφορά για τη χρήση αντιβιωτικών γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί αυτό γιατί είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ Συμφωνώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ήταν ε, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης ενός ε, ε, νομοθετικού προτύπου για την καλή μεταχείριση και ευημερία των ζώων, που ωστόσο δεν είμαστε σε θέση να διαδώσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, ένα λεπτό, παρακαλώ. Έχουμε ένα πρόβλημα με την αγγλική μετάφραση, μια στιγμή λέει κύριε Καπούτο. Λοιπόν, το ίδιο βλέπουμε και στην περίπτωση των σφαγίων και της σφαγής. Οι προϋποθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφορούν μόνο την ε, εσωτερική αγορά και όχι τα εισαγόμενα προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε μια παγκόσμια στρατηγική και να ακολουθήσουμε τους ε, κανόνες της παγκόσμιας οργάνωσης για την ευζοία ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει αυτό να, αποτελεί, να οδηγεί μάλλον σε ένα συγκριτικό μειονέκτημα λόγω ε, αυξημένου κόστου ή πιο περίπλοκων διαδικασιών στο εξωτερικό στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν στρεβλώσει που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με τι διαφορέ ε, που έχουν να κάνουν με την ευημερία των ζώων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των κανόνων που ισχύουν εκτό αυτή, ειδικά για τα αυγά και τα προϊόντα βάση αυγών και εκείνα τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με βόλιο κρέας. Οι μακροβιολογικές εξετάσεις, ειδικά για τα προϊόντα κρέατος που έρχονται από, βόδι, από βόλιο κρέας, αποδεικνύουν για εκείνα τα προϊόντα που προέρχονται από τη Βραζιλία ότι δεν τηρούνται οι κανόνες και μάλιστα γίνεται και παραποίηση πιστοποιητικών για να εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρέας που έχει και ηλικία ανά των 10 ετών. Μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να μας ενημερώσει για όλους τους ελέγχους που έχουν γίνει και τα ευρήματά τους, ειδικά όσον αφορά με την ε, ε, Βραζιλία και τις σχετικές προσαρμογές της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ, αφού μας είπατε κι εσείς ότι προχωρείτε σε μια προσαρμογή και υλοποίηση των κανόνων αυτών. Αφού χρησιμοποιήσετε εσείς οι ίδιοι αυτόν τον όρο, μπορείτε να μας πείτε τι κάνετε ακριβώς. Ευχαριστώ, Χάσελκαμπ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Με χαρά ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ε, σημαντική την προστασία των ζώων. Αλλά επί της ουσίας δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Πολλά λόγια και λίγα έργα. Και από την έκθεσή σας δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Επίσης βλέπουμε ότι μπορεί να έχουν γίνει κάποια μικρά βήματα για την ε, καλή μεταχείριση των ζώων, όπως σε παραδείγμα το να μην κρατούνται σε κλουβιά αλλά αυτά είναι δεκαετία του 90 και εντωμεταξύ δεν έχει προχωρήσει τίποτε. Φαίνεται ότι οι φιλοδοξίες οι μεγάλες που είχαμε για την προστασία των ζώων έχουν εξανεμιστεί. Ή πάντως δεν τηρούνται οι κανόνες. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να μας λέτε ότι αυτοί οι κανόνες για την προστασία των ζώων, αυτοί οι κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να φέρουν κάποιες αλλαγές και σε παγκόσμιο επίπεδο για την ε, προστασία των ζώων. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το εμπόριο δεν προσβλέπει καμία συμφωνία για προστασία ζώων και η συμφωνία με την Ουκρανία παραδείγματι επίσης δεν κάνει λόγο γι' αυτό. Το ελεύθερο εμπόριο, και αυτό είναι το χειρότερο παράδειγμα που μπορούμε να προβάλλουμε, είναι αυτό που έχει να κάνει με τη μεταφορά των ζώων όπου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ισχύουν οι κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι κάποιες προϋποθέσεις ισχύουν ε, για την μεταφορά ζώων και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχουμε δύο φορές επισημάνει ότι δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες για την προστασία των ζώων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν οι μεταφορεί των ζώων ότι οφείλουν να τηρούν αυτού του κανόνε στη μεταφορά. Μπορείτε να μα δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα λοιπόν. Ποιοι είναι οι κανόνε οι οποίοι τηρούνται και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο εντό. Ο κύριο Αντριού. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ε, έκθεση καταρχάς, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση, αλλά και για τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού. Θα να σας παρακαλέσω κι εγώ να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με την τήρηση των κανόνων για την ανταγωνιστικό, και την ανταγωνιστικότητα. Με την παγκοσμιοποίηση βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πώς αναπτύσσεται το γεωργικό μοντέλο. Επομένω, οι οικονομικοί όροι έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε και στα, ε, στη χρήση των αντιβιωτικών αλλά και στα μέσα φυτοπροστασίας που χρησιμοποιούνται στις μεγάλες ιδίω εκμεταλλεύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν έχετε ε, μελετήσει τη συμπεριφορά του καταναλωτή και εδώ ιδιαιτέρως εάν υπάρχουν καταναλωτές, όπως είναι οι vegan που είναι όλο και πιο πολύ άριθμοι πλέον, εκείνοι που τρώνε μόνο φυτικά προϊόντα και κανένα προϊόν ζωικής προέλευσης, και αν αυτοί μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο παραγωγής, γιατί βέβαια είναι το τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας της κατανάλωσης. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Βουαζού. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, όταν μιλούμε για ε, ευημερία των ζώων πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Καταρχάς θα πρέπει να κοιτάξουμε για το θέμα της, ε, σήμαν, της επισήμανσης η οποία επιβαρύνει ιδιαίτερα οικονομικά τον ε, παραγωγό, ειδικά αυτόν ο οποίος θέλει να είναι τυπικός. Και βεβαίω είναι ο καταναλωτή απαιτητικό ω προ την ευημερία των ζώων, ω προ την προέλευση των προϊόντων. Είναι διατεθειμένο να καταβάλει ψηλότερο τίμημα προκειμένου να έχει μια ανιχνεύσιμη προέλευση. Πρέπει λοιπόν να προσανατολιστούμε και να υπερασπιστούμε εμείς ως νομοθέτες την ε, ευάρετη ε, ενάρετη μάλλον παραγωγή ε, και βεβαίως να προστατεύσουμε τη δική μας παραγωγή σε σχέση με τα προϊόντα που έρχονται από, ε, από τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς να σέβονται τους ίδιους κανόνες. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει και να επιβαρύνουμε περιβολικά τον παραγωγό. Φερρυπίν, μεταφορές των ζώων. Εδώ πέρα νομίζω σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Επίσης η παραδοσιακή τελετουργική σφαγή χαλάλ, για την οποία δεν είπατε κουβέντα εσείς κυρία μου, και όμως έχει οπωσδήποτε ε, τεράστια σημασία εάν θέλουμε να μιλάμε για την καλή μεταχείριση των ζώων. Ευχαριστώ κύριο Σάγνιου. Ευχαριστώ πολύ. Ενδιαφέρον εδώ στην έκθεση ήταν ότι μας είπε ότι Μπορεί οι τρίτες χώρες να τηρούν ε, και τις δικές μας προδιαγραφές, αλλά είναι, παραμένουν αυτές ανταγωνιστικές γιατί έχουν πιο φτηνό ε, μισθολογικό κόστος. Άρα λοιπόν έχουμε προβλήματα και έχουμε πρόβλημα γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι τρίτων χωρών. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν τρεις σε εκκρεμότητα ε, οχλήσεις για χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν τηρούν τους κανόνες για, την, ε, για τους τάβλους. Επίσης όλη αυτή η ιστορία και τα εύκολα λόγια που ε, ξοδεύεται για να καθησυχάσετε τον κόσμο ότι έρχεται η αύξηση θερμοκρασίας του πλανήτη που τα έχει προξενήσει ο άνθρωπος και άρα θα ε, είναι πιο ήπιοι χειμώνας, το βλέπουμε αυτό το Μάρτιο που είναι παγωμένο συνέχεια. Ε, αυτό όμω έχει συνέπειε και σε σχέση με τη συμπεριφορά του καταναλωτή στα, ζώια, ε, στα ζωικά προϊόντα. Αυτό που θα έλεγα λοιπόν εγώ είναι κοιτάξτε τι κάνετε εσείς, ε, κοιτάξτε τα του οίκου σας και αφήστε τους άλλους να τα τα δικά τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ. Βεβαίω, όλοι υποστηρίζουμε την καλή μεταχείριση των ζώων, αλλά δεν μα είπατε με ποιο τρόπο υπολογίζετε το κόστο παραγωγή των προδιαγραφών που θέλετε να επιβάλλετε. Διότι αυτό θα κρυθεί, πιστεύω, από την στρέβλωση, και το έχουν πει πολύ πριν από μένα, των τιμών σε σχέση, το, και του ανταγωνισμού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρε εκτό αυτή, ιδιαίτερω δε τη Βραζιλία αλλά και γενικότερα τη Μερκοσούρ στο πλαίσιο αυτού του ανταγωνισμού. Ε, πώς λοιπόν διερευνά τις ε, ενισχύσεις που μπορεί να λαμβάνουν η σχετική παραγωγή, έτσι ώστε να στρεβλώνουν τελικά τον ανταγωνισμό, τους όρους και το κόστος ε, χρηματοδότησης στη Βραζιλία, αλλά γενικότερα στην, στο Μερκοσούρ, είναι πολύ χειρότερες συνθήκες διαβίωση των ζώων. Δεν καταγγέλλονται όμως από τις οργανώσει για την προστασία των ζώων και παρόλα αυτά επιτρέπεται να εισάγονται τα προϊόντα αυτά. Εδώ ο κύριος Χόισλιν έχει το λόγο. Κύριε εκπρόσωπε της Επιτροπής, ε, μας δώσατε μια θετική εικόνα του τρόπου με τον οποίο συνεχίσει τι προσπαθίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν είναι σε θέση να επιβάλλει ομοιόμορφε προδιαγραφέ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είδαμε εξαιρέσει, παρεκκλήσει από τη Γερμανία, αλλά και άλλες, προ όφελο μάλλον τη Γερμανία, αλλά και άλλες χώρες. Και άρα δεν βλέπουμε να ισχύει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Καταρχά λοιπόν πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ε, με τον ίδιο τρόπο η νομοθεσία για την προστασία των ζώων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά κοιτάξουμε και έξω. Και επίση τον έλεγχο στι μεταφορέ ζώων βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικέ ποιότητε ελέγχων με πολύ διαφορετικά αποτελέσματα και ευρήματα, πως θα έπρεπε να τυποποιηθούν κατά κάποιο τρόπο οι διαδικασίες ελέγχου, διότι εδώ σημειώνονται πολύ μεγάλα κενά, και το είπαν και πολλοί άλλοι, ε, νωρίτερα στο εμπόριο εκτός, στη διακίνηση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα ήταν καλό να κοιτάξουμε και αυτή τη διάσταση. Πολλά έχουμε τόσο άλλο να κάνουμε, πολλά θα μας απασχολήσουν στο διεθνές μας εμπόριο. Καλό θα ήταν λοιπόν να τηρηθούν αυτές οι προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού, ούτως ή άλλως να επιμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, γιατί βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν... ε, ε συστήματα εκτροφής ε, των ζώων που δεν τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αντιστοιχούν σε κανένα ως τύπου προδιαγραφές. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα έλεγα να είμαστε λίγο πιο επικριτικοί και ας προσπαθούμε τις δικές μας καλές προδιαγραφές να τις εξάγουμε και προς τα έξω. Έχουμε πολλά ακόμα να εξασφαλίσουμε και επίσης θέλω να ρωτήσω γιατί δεν έχει γίνει τίποτα σε σχέση με τις... Ε, ε, με την εκτροφή των ε, κουνελιών ε, κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα κάνω την εισαγωγή που σκόπευα ο κύριος Βάιτς, γιατί ο κύριος Χόισλινγκ με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό. Μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχουν οι Ευρωπαίοι παραγωγή Ε, δεν έχουν μάλλον η παραγωγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μειονέκτημα, μάλλον πλέον έκτημα σε σχέση και με τις συνθήκες ε, εκτροφής των ζώων. Αλλά θα ήθελα να πω, μια και αναφέρθηκε και νωρίτερα η Ουκρανία, αλλά και άλλες χώρες, πώς προβάλλουμε το πλεονέκτημά μας ε, το ανταγωνιστικό σε σχέση με χώρες οι οποίες δεν τηρούν τις ίδιες προγραφές. Πώς θα το εξηγήσουμε αυτό στο γεωργό μας. Και πώς επιτρέπουμε να γίνονται εισαγωγές κρέατος, γάλακτος, αυγών που δεν τηρούν τις ίδιες αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές γιατί αν είναι έτσι οι δικοί μας παραγωγοί δεν έχουν καμιά ελπίδα επιβίωση ούτε καν μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο κύριος Γιάρ έχει, κύριε Γιάρ. Ναι, κατέκλεισε ο ενθουσιασμός γιατί ο συνάδελφός μου τα είπε τόσο ωραία που ήθελα να το επισημάνω, το έχει δίκιο. Ναι, λοιπόν, είπαμε ότι πρέπει να μεριμνήσουμε για παγκόσμιες προδιαγραφές, μια χρυσή γέφυρα θα λέγαμε, Golden Bridge. Θα μας βοηθούσε, θα έλυνε όλα τα προβλήματα, να έχουν όλοι τις ίδιες προδιαγραφές, τις ίδιες συνθήκες, να αγωνιστεί λοιπόν ακόμη και να συνεχίσει να αγωνίζεται για προδιαγραφές σε επίπεδο παγκόσμιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά μια και ο κόσμος δεν είναι ιδεώδης και κάπου υπάρχουν διαφορετικέ προδιαγραφέ, κάπου είναι καλύτερα, κάπου είναι χειρότερα τα πράγματα σημειώνονται ως αποτέλεσμα και διαφορετικό κόστος και στρεβλώσεις ανταγωνισμού. Έτσι λοιπόν ναι, μπορεί να υπάρχουν ε, και έχει δίκιο εδώ ο συνάδελφος ε, στρεβλώσεις οι οποίες μας ενοχλούν. Ε, πρώτον όταν εξάγουμε τρίτα κράτη μπορεί βεβαίως λίγα ζώα να εξάγουμε εμείς σε τρίτα κράτη αλλά πάλι ως Ευρωπαϊκή Ένωση φέρουμε ευθύνη Μέχρι την ώρα της κατεργασίας του υλικού προϊόντος δεν μπορούμε να πούμε πέρασε ε, τα σύνορά μας ε, το προϊόν και δεν μας απασχολεί πλέον τι γίνεται. Ε, ε, πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τον τρόπο μεταφοράς των ζώων, τα, υπάρχουν ίδιες προδιαγραφές στη σφαγή κτλ. Και το άλλο το οποίο περισσότερο ακόμη αφορά και το ανέφερε και ο συνάδελφος νωρίτερα για τι εισαγωγέ, γιατί βεβαίως τεχνικές προδιαγραφέ, είναι πολύ σημαντικές. Εάν πρέπει να έχει ο Σολίνας μια ετικέτα μπλε, ξέρω εγώ, ναι εντάξει, δεν μπορεί να έρθει κανείς και να βάλει μια κόκκινη ετικέτα. Πολύ ωραία, αλλά η εφημερία των ζώων δεν είναι τεχνικές προδιαγραφέ μόνο. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εις βάρος των δικών μας παραγωγών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μεριμνούμε ώστε τα εισαγόμενα προϊόντα να πληρούν απολύτως και να τιμούν τις ίδιες, τεχνι... τις ίδιες ε, προδιαγραφές που ισχύουν στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν πρέπει και προς τα έσω αλλά και προς τα έξω να το σε αγωγές και εξαγωγές και κάτι ακόμη που ίσως να μην ενδιαφέρει πολύ με την έννοια ότι είναι χαμηλό το κόστος, ε, η επιβάρυνση του κόστους. Ε, είναι το εξή ότι το μικρό μειονέκτημα το οποίο μπορεί να παρουσιάζεται εδώ ή να αναλύεται εδώ μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη στρεβλώση. Ευχαριστώ και είναι δική μας ευθύνη. Μπούντα. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Είμαι αρκετά διστακτικός ό,τι φορά κάποια πράγματα που ακούστηκαν στην παρουσίαση της έκθεσης. Είπατε για το κλίμα, το που μπορεί να επηρεάσει, την παραγωγή ε, χειρίου κρέατος ή πουλερικών. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα προδιαγραφές όμως. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μιλήσω για την ανταγωνιστικότητα. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταλαβαίνει ότι χαμηλώνοντας τα πρότυπα ποιότητας ε, κατά την εισαγωγή προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δημιουργούμε ε, μια κατάσταση εξαιρετικά άνηση όπου η παραγωγή μας είναι σε θέση και μπορεί να χρεοκοπήσουν τι να πω δεν μπορεί να, να συγκριθεί το κόστος στο Μερκοσούρ με το κόστος εδώ. Είναι διαφορετικά τα πρότυπα ποιότητας και αφήνουμε προϊόντα να προέρχονται από διάφορες περιοχές του κόσμου να εισάγονται που δεν πληρούν τις προδιαγραφές μας. Οπότε δημιουργούμε συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού και αυτό είναι επιβλαβές για τους παραγωγούς μας. Θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ε, επιβίωσή τους. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε το ζήτημα σφαιρικά. Υπάρχουν διάφορες πτυχές. Ε, ε, τα αντιβιωτικά, ε, οι ζωοτροφές, φάρμακα. Εμείς έχουμε πολύ αυστηρούς κανόνες εδώ και πολύ αυστηρή εποπτεία επίσης εφαρμογής των κανόνων. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μας δώσετε μια ανάλυση από διεθνή προοπτική ε, που θα μπορούσε να, να, να περιγραφεί ως soft power ε, ότι δίνουμε το παράδειγμα, ε, ότι ευαισθητοποιούμε, όμως υπάρχει και κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, το θέμα του εμπορίου και είναι πολύ ασαφής η επιρροή που έχει στις εμπορικές συμφωνίες το θέμα της μεταχείρισης των ζώων. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι κανόνες ε, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου, τους οποίους ε, ακολουθεί η Κομισιόν στις συμφωνίες της. Ε, εξαρτάται από τη μία συμφωνία στην άλλη. Ε, δεν μπορεί να είναι ουσια... ή, ή μπορεί να είναι ουσιαστικό μέρος μιας εμπορικής συμφωνίας το θέμα της μεταχείρισης των ζώων ή όχι. Πότε θα κινητοποιηθεί η η μπορει να ειναι ουσιαστικο μερος μιας εμπορικης συμφωνιας στο θεμα της Επιτροπή ε, για να θεσπίσει κάποια πρότυπα, να τα επιβάλλει και μετά να περιμένει βεβαίως και τις προσφυγές που θα υπάρξουν. Γιατί με προσφυγές λειτουργεί ο ΠΟΕ. Δεν λειτουργεί έτσι ο κόσμος του ΠΟΕ. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο γενναίοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πιο γενναία. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η σχέση μεταξύ των εμπορικών συμφωνιών και της ευημερίας των ζώων. Και βεβαίω ε, συμφωνώστε με την ανάλυση σα. Είναι σημαντικό να καταλάβουν τα μέλη αυτό που λέτε, ότι, ε, είναι, ότι η ευημερία των ζώων δεν είναι ένα κόστος ε, σημαντικό για την παραγωγή. Αλλά τα στοιχεία που αφορούν την ευημερία των ζώων μπορεί να μην έχουν τόσο μεγάλη διαφορά στο κόστος, αλλά είναι ένα θέμα αρχής για μας. Εφόσον ζητούμε από του γεωργού μα να δεσμεύονται από αυτού του κανόνε, θα πρέπει να πω στου ίδιου κανόνε ε, αυτοί που εξάγουν προϊόντα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει αυτό να το αναφέρει η Κομισιόν και να το προωθήσει. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όπως και οι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι βεβαίω είναι τα μηνύματα θετικά όπως μας παρουσιάζονται, αλλά θα ήθελα να ήξερα πόσα κράτη συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα εάν επί παραδείγματι συμπεριελήφθη η Τουρκία ή, μία, ή άλλα, μη, ε, μέλη της, ή άλλα κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν τηρούνται οι ίδιες προδιαγραφές ε, μέσα στην Ευρώπη από ό,τι διαπιστώνουμε φαντάσου εκτός Ευρώπης τη ισχύει. Θέλουμε ιδιαίτερος για τη σφαγή αλλά και για τις μεταφορές των ζώων, για τη μεταφορά των ζώων να ξέρουμε και βεβαίως πόσα είναι τα ζώα τα οποία ζωντανά εξάγονται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να φέρουν αποτελέσματα οι έλεγχοι ουσιαστικά και δεν αρκεί να βλέπουμε οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές και να μην εφαρμόζονται. Από ό,τι φαίνεται η Βουλγαρική ε, Προεδρία δεν έχει ιδέα Ποιο πρέπει να κάνει του ελέγχου, ε, πότε παραπέμπει στον ένα, πότε στον άλλον. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο απαιτητικοί για το τι ισχύει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτό αυτή, ιδιαίτερα για τα ζώα τα οποία πηγαίνουν για σφαγή, μεταφορά του και, ωραί, και προϋποθέσεις σφαγής. Και αν δεν αρκούν ε, οι κανόνε, πρέπει να του επεξεργαστούμε και να τους βελτιώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζουάνα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ συζητούμε τους ε, κανόνες της διατάξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίους και επιβάλλουμε στους ε, παραγωγούς. Καλό είναι αυτό σε έναν βαθμό, διότι μας ε, επιτρέπει να βελτιώσουμε την προστασία των ζώων, αλλά και τις υγείας του καταναλωτή. Εγώ όμως ρωτώ αυτοί οι κανόνες ισχύουν για τρίτες χώρες, εφαρμόζονται από τους εξαγωγούς, εξαγωγείς, ζωικών προϊόντων στην Ευρώπη. Υποχρεούνται αυτοί να ε, τηρούν τους ε, κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων. Υπάρχουν ε, κανόνες που έχουν αποδεχθεί και τρίτες χώρες και μπορούμε να εξακριβώσουμε ότι όντως τηρούν αυτοί οι εξαγωγείς τους ίδιους κανόνες που έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης υπάρχουν τρόποι μέτρησης υπολογισμού, μονάδες μέτρησης, βιολογική, ε, δείκτες, ε, ε, τεχνικά χαρακτηριστικά, εν που να μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Υπάρχουν συνθήκες λοιπές πριν, τις, ε, πριν των σχετικών με την ε, εκτροφή των ζώων, ε, όρια εργασίας, συνθήκες εργασίας, υγεία και υγιεινή στο χώρο εργασίας που τηρούνται και στις άλλες χώρες για να μπορούμε να συγκρίνουμε. Γιατί βεβαίως αναγνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να από περιοχή σε περιοχή. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο το τι, σημαίνει, τι συμβαίνει στο, σε τοπικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Μαγκίνες, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πολλά ζητήματα που με απασχολούν τα έθιξαν άλλοι συναδελφοί. Εγώ λοιπόν θα περιοριστώ σε ένα συναφές ε, ε, σχόλιο γιατί θεωρώ ότι θα μας παρακολουθούν αρκετοί πολίτες και πολύ συχνά μας λένε οι γεωργοί που συναντώ εγώ τουλάχιστον στην εκλογική μου περιφέρεια, ότι οι άνθρωποι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πολύ ασχολείται με τα ζώα παρά με τους ανθρώπους. Ε, σε περιόδους όπως η τωρινή ε, χειμερινή περίοδος που έχει δει τεράστιες καταστροφέ, ε, καταστροφές, καταιγίδες, ε, χιόνι κτλ, χιονοθύλες, πρέπει να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι μεριμνούμε και για τον άνθρωπο, για τον γεωργό, για την οικογένειά του, που υφίσταται μεγάλες πιέσεις σε μια περίοδο που γεννούν και όλα στα ζώα, που έχουν τα μικρά αρνιά και πρέπει να είναι σε θέση να τα ε, προστατέψουν, να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Έτσι λοιπόν όταν πολλές φορές λέμε μέσα σε αυτές τις αίθουσες που συνεδριάζουμε ότι α, πρέπει να επιβάλλουμε συνθήκες ε, παραγωγής κτλ δίνουμε την εντύπωση ότι δεν μεριμνούμε αρκετά, ότι δεν έχουμε στο μυαλό μας τον παραγωγό όπως θα έπρεπε και την οικογένειά του. Οπότε ας κοιτάμε πάντα, με ό,τι συζητάμε, ότι απευθυνόμαστε σε κάποιους ανθρώπους που υφίστανται τεράστια πίεση. Πρέπει να τους δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό και να δράσουμε αναλόγως. Και να αναγνωρίσουμε βεβαίως τη δουλειά. Μάλιστα. Ακούσαμε όλους τους συγκεκριμένους στο κατάλογο των αγορητών. Θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Σκριβάνο, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να απαντήσει σε ερωτήσεις ε, και στα προβλήματα που επισήμαναν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω βεβαίως, ε, να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στην εφαρμογή, στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας κάτι που δεν αποτελούσε μέρος ε, του πεδίου έρευνας αυτής της έκθεσης. Ε, αυτό που θέλω βεβαίως εγώ να σας πω είναι ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια από τις βασικές προτεραιότητες ε, είναι να εγγυηθούμε την εφαρμογή της υπάρχουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και ένα από τα ζητήματα στο, στα οποία δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση είναι το θέμα της μεταφοράς ζώντων των ζώων, το ανέφεραν κάποιοι από εσάς, υπάρχει μια διεύθυνση στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ που διενεργεί ελέγχους στα κράτη-μέλη, αποστολές ε, και σε χώρες όπως η Τουρκία για να αξιολογηθεί η κατάσταση ε, και να παρακολουθούμε το θέμα των μεταφορών. Υπάρχουν και άλλες ε, δραστηριότητες υπό την αιγύδα της Κομισιόν συνάντηση των εθνικών σημείων επαφής για τις μεταφορές. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας ε, για την Ευημερία των Ζώων έχουμε δημιουργήσει μια υποομάδα για τις μεταφορές. Το παίρνουμε λοιπόν πολύ στα σοβαρά το ζήτημα και έχουμε απόλυτη συνέστηση της σημασίας ε, των συνθήκων ε, που θα πρέπει να πληρούνται, των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται ε, για τη μεταφορά ε, ζών των ζώων και προς τρίτες χώρες. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα βεβαίως για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Εμείς ε, όμως ελέγχουμε αυτή την εφαρμογή. Επίσης, ε, τέθηκαν μια σειρά από ερωτήματα σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη μελέτη αυτή. Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο ε, στην ανταγωνιστικότητα των μέτρων για την ευημερία των ζώων. Ε, βασιζόμαστε σε τέσσερις πηγές πληροφορίας. Η, η υπάρχουσα βιβλιογραφία, ε, ή συνεντεύξεις με διάφορες ενώσεις επιχειρήσεων ή εμπορικές ροές και δύο εστιασμένες μελέτες ε, ε, σε κτηνοτρόφους εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επιλογή ε, σε χώρες Ουκρανία, Λίβανος, Χιλή, Βραζιλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ταϊλάνδη, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Νέα Ζηλανδία, και Αυστραλία. Αυτές είναι οι 12 χώρες που απάντησαν ε, στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, εκτός από την Ταϊλάνδη και την Νέα Ζηλανδία που δεν απάντησαν. Ε, αυτά σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δυνατότητα στη μελέτη αυτή ε, να έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα καινοτομία την επιλογή των καταναλωτών είναι κάτι το οποίο ανέφεραν κάποιοι από εσά. Ε, δεν κατέστη εφικτό να έχουμε δεδομένα που να, δείχνει, που να δείχνουν ποια είναι η συνεισφορά σε ό,τι αφορά την ε, εφημερία των ζώων. Διότι συχνά αυτό συνδέεται με άλλα ζητήματα. Ε, μπορεί να συνδέεται σε, στη βιολογική παραγωγή, σε προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Είναι δύσκολο να προσμετρήσουμε το θέμα της ευημερίας των ζώων σε ό,τι αφορά την επιλογή των καταναλωτών. Δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτό ε, και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να καλύψουμε το ζήτημα αυτό. Επίσης, πολλοί από εσά αναφέρθηκαν σε ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές. Να υπενθυμίσω ότι ως μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε ε, τις δεσμεύσεις μας. Ε, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τα πρότυπά μας σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό και ο αντίκτυπος ε, αποτυπώνεται μέσω της βελτιωμένης συνεργασίας. Πριν από μερικά χρόνια όταν αρχίσαμε τις διπλωματεύσεις με τρίτες χώρες ε, στα πλαίσια εμπορικών ε, συμφωνιών ήταν αδύνατον να, να συμπεριλάβουμε ε, το θέμα αυτό ούτε καν στη μέση διάταξη ενώ τώρα υπάρχουν χώρες που μας ζητούν την υποστήριξή μας για να βελτιωθούν οι συνθήκες σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση των ζώων. Το να βάλουμε το θέμα της ευμερίας των ζώων λοιπόν ε, στην διεθνή σκηνή σημαίνει η ανάπτυξη διεθνών προτύπων στα πλαίσια του ΟΑΗ. Αν θέλουμε τα πρότυπα αυτά να εφαρμοστούν παγκοσμίως θα πρέπει όμως να τα δεχτούν και οι άλλοι. Γι' αυτό η Κομισιόν συστηματικά περιλαμβάνει διατάξεις περί ευημερία των ζώων, με έναν άλλο, τον άλλο τρόπο στις συμφωνίες με τρίτες χώρε, ε, με τι οποίε οποίες πραγματευόμαστε Από τότε που έχουμε λάβει βεβαίω τη σχετική εντολή από το Συμβούλιο, σε κάθε συμφωνία, σε κάθε μνημόνιο ε, εμπορικό υπάρχει το θέμα της ευημερίας των ζώων, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες ε, σε πολλές χώρες για το ζήτημα αυτό. σε ό,τι αφορά τώρα το πώς συνδέεται αυτό με την ε, αντίσταση, την αντιμικροβιακή, αυτό δεν έχει σχέση με την έκθεση, αλλά το θέμα αυτό ε, είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, εργαζόμαστε ενεργά λοιπόν στα πλαίσια του ΟΑΗ και άλλων διεθνών οργανισμών για να το αντιμετωπίσουμε. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες διατάξεις που έχουν να κάνουν με την επισήμανση ιδιαίτερα για τα ε, αυγά. Εξετάζουμε το θέμα των διεθνών προτύπων και πώς εφαρμόζεται, διότι ήταν τα πρώτα πρότυπα που είχε εγκρίνει ο ΟΑΗ, αυτά που αφορούν την σφαγή και τη μεταφορά. Ελπίζω να απάντησα στα ερωτήματά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την απάντηση στις ερωτήσεις. Φαντάζομαι ότι έχετε επίγνωση ότι υιοθετούμε μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση στην Επιτροπή μας για την καλή μεταχείριση των ζώων. Ενώ σε άλλες επιτροπές, ονόματα δεν λέμε, ε, τέτοιου είδους ζητήματα είναι ακόμη πιο επίμαχα. Εμείς είμαστε πιο προσγειωμένοι, πιο ρεαλιστικοί στην προσέγγιση μας για την καλή μεταχείριση των ζώων. Βέβαια, Είμαστε όλοι υπέρμαχοι της ε, κοινοτικής νομοθεσίας και των προδιαγραφών μας ε, για την καλή μεταχείριση των ζώων. Βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε πώς επηρεάζουν αυτές οι προδιαγραφές και διατάξεις την ανταγωνιστικότητά μας και να μην την περιορίζουν. Γιατί έχουμε καλούς στόχους, ε, αλλά θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε να εφαρμόζονται ομοιόμορφα στα κράτη-μέλη. Γιατί μερικές φορές συνειδητά η παραγωγή δεν εφαρμόζουν όλες τις προδιαγραφές και πρότυπα, προσπαθώντας να μειώσει το κόστος παραγωγής. Γιατί το κόστος είναι σημαντικός παράγοντας. Και Τελικά όμως μερικές φορές η παραβίαση των κανόνων και των προδιαγραφών γυρίζει μπούμεραγκ ει βάρο των παραγωγών. Θα πρέπει και αυτό να το λάβουν υπόψη. Ευχαριστώ θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό κάποια στιγμή. Γιατί το θέμα της καλής μεταχείρισης ε, των ζώων στη μεταφορά θα μας απασχολήσει και αργότερα στη συνεδρίαση των συντονιστών. Ε, θα το εξετάσουμε γιατί ε, υπευλήθη έτοιμα για σύσταση ειδική επιτροπής ε, για να αγγίψει αυτό το θέμα της ε, μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά. Και η κυρία Μίλλερ ασχολείται ιδιαίτερως με το θέμα αυτό, οπότε σίγουρα μας ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα και από θέμα καλής μεταχείρισης αλλά και από οικονομικής απόψεως. Σας ευχαριστώ θερμά ε, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ήρθε στην Επιτροπή. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο 6 δηλαδή. Κοιτάω προς την κυρία Αγγιλέρα που είναι η αρμόδια για το θέμα της Παρασκευής, διάθεση στην αγορά και χρήσης φαρμακούχων ζωοτροφών, καθώς και την κατάργηση της οδηγίας 90-167 του Συμβουλίου. Ήδη ε, στην προηγούμενη συζήτηση επισημάθηκα κάποια προβλήματα σε σχέση με τα αντιβιωτικά, τη χρήση των ε, φαρμάκων στις ζωοτροφές. Αλλά νομίζω ότι πλέον κατάλληλη να μας ενημερώσει για το θέμα αυτό είναι η συγγήτρια η κυρία Αγγιλέρα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ε, για την κατάσταση των συζητήσεων σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Ε, είχαμε μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη των τριμερών διαλόγων και μάλιστα αδικαιολόγητη δεν ε, εξηγείται από τον κανονισμό. Αλλά η εντολή που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον κανονισμό αυτό συνδέεται άμεσα, αναπόσπαστα, με τις συζητήσεις που γίνονται στον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Η αρμόδια επιτροπή για τον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και ε, εκεί καθυστέρησε πολύ το Συμβούλιο στη Συμφωνία. Και παρόλο που έχουμε εγκρίνει το θέμα εδώ και πολύ καιρό, οι τριμερεί ε, διάλογοι για τις φαρμακούχε ζωοτροφέ άρχισαν πολύ πρόσφατα, με μεγάλη καθυστέρηση. Ο πρώτος τριμερή διάλογο έγινε σε 6 Μαρτίου. Νομίζω ότι ήταν θετική η έκβαση του πρώτου τριμέρους διαλόγου. Είχε γίνει μια τεχνική άλλωστε προεργασία πριν την διεξαγωγή του πρώτου τριμέρους διαλόγου. Ο Γκονσάλο, η Γραμματεία, η Μαγδαλένα, οι συνεργάτες μου και άλλοι τεχνικοί συνεργάτες και σύμβουλοι και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έκαναν πολύ σημαντική τεχνική προεργασία και προλύαναν το έδαφος για τον τριμέρι διάλογο, οπότε στις 6 Μαρτίου στον πρώτο τριμερή διάλογο σημειώσαμε αρκετή πρόοδο σε πολλά σημεία θα έλεγα σε ό,τι αφορά μερικά άρθρα καθώς και τα παραρτήματα. Το πρόβλημα στη συζήτηση του κανονισμού αυτού στον τριμερή διάλογο είναι ακριβώς επειδή συνδέεται αναπόσπαστα με τον άλλο κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα, στα θέματα των ορισμών για παράδειγμα ή σε μερικά άλλα ζητήματα. Ακριβώς ε, λόγω της αλληλεπίδρασης των δύο κανονισμών Προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις συμφωνίες στον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα, γιατί πολλά άρθρα εκείνου του κανονισμού θα επηρεάσουν και το δικό μας κανονισμό για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Οπότε, σε 6 Μαρτίου ήδη καταλήξαμε στη συμφωνία για σημαντικά θέματα, σχεδόν ε, διεκπαιρεώσαμε το 50% και κάτι των ζητημάτων των εκκρεμωτήτων και τον, ο επόμενος διάλογος θα γίνει στις 26 Απριλίου. Προσωρινά αυτό προγραμματίσαμε. Οπότε, η κυρία Γκροστέτ που είναι αρμόδια για τα κτηνιατρικά φάρμακα ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, προωθήσει το θέμα και έχουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε και εμείς στο δεύτερο τριμερή διάλογο θα γίνει όπως έχουμε προγραμματίσει στις 26 Απριλίου. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των συζητήσεων για τα κτηνιατρικά φάρμακα, για την έκθεση Γκροστέτ. Αλλιώ θα πρέπει να αναβάλουμε κι εμεί τον τριμερή διάλογο για άλλη στιγμή. Αν θέλετε μπορώ να επισέλθω και σε συγκεκριμένα θέματα. Πάντω ήδη στον πρώτο τριμερή διάλογο σημειώσαμε εντυπωσιακή πρόοδο με το Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο έχουμε κάποια σύμπτωση απόψεων σε αρκετά θέματα και επίσης στον επόμενο τριμερή διάλογο που ελπίζω ότι θα γίνει τελικά στις 26 Απριλίου, αν δεν αναβληθεί, να διατρανώσουμε και πάλι την βούλησή μας, τη δική μου και των άλλων σκιωδών εισηγητών, να καταλήξουμε σε σωστές διατάξεις για την παρασκευή των φαρμακοχών ζωοτροφών, αλλά και για τον άλλο τρόπο χορήγησης ε, κτηνιατρικής ε, αγωγής ε, στα φάρμακα όπως είναι με τα διαλυτά φάρμακα είτε με την επίπαση στη ζωοτροφή. Γιατί ήδη έχουμε ε, κάποια ε, στοιχεία που θα πρέπει να, αποσαφηνίσουμε. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα αντιβιωτικά, τη χρήση των αντιβιωτικών, που φυσικά επηρεάζει και ζώα και ανθρώπους και η ευθύνη δική μας στους τριμερείς διαλόγους είναι να θεσπίσουμε μια καλή νομοθεσία για τα επόμενα χρόνια, ώστε η υγεία των ζώων να ελέγχεται δεόντως και να προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ε, λαμβάνοντας υπόψη και το πρόβλημα που έχουμε με τα αντιβιωτικά και τη μικροβιακή αντοχή. Ευχαριστώ θερμά τους και ηγητές φυσικά για την αγαστή συνεργασία που έχουμε μέχρι στιγμής και που ευελπιστώ ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Και να πω ότι είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα, πολύ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κοιτώ εδώ την ομίγυρη. Θέλει κανείς το λόγο για να υποβάλει ερωτήσεις προς την κυρία Γιλέρα. Θέλετε, έχετε απορίες, θέλετε να μάθετε κάτι. Κύριε Μπούντα, δεν έχουμε και πολύ χρόνο και δεν έχουμε και πολλά να πούμε. κύριος Μπούντα. Ναι, όχι ακριβώς ερώτηση. Επειδή είχα συμμετάσχει ως σκιώδης εισηγητής ε, σε σχέση με αυτούς που προτείνουν ε, να δίνονται αυτές οι ε, οδηγίες γιατί επί παραδείγματο στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει δυνατότητα τη συνταγή, δεν υπάρχουν αρκετοί κτηνοτρόφοι, να την εκδίδουν άλλε αρχέ. Ε, μήπως μπαίνουμε σε κάποια επικίνδυνα παιδεία. Κάτι τέτοιο ισχύει και στην Ρουμανία λίγο πολύ. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν είναι κτηνοτρόφοι απαραίτητοι, κτηνίατροι απαραίτητα, ε, αλλά έχουν περάσει από μια κτηνιατρική σχολή, μπορούν να εκδίδουν συνταγές. Είναι δυνατόν έτσι να γίνεται η σταγογράφηση των αντιβιωτικών. Επίσης νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε να μην δοθεί από άλλα κράτη-μέλη τέτοιου είδου άδεια σε μη κτηνιάτρους. Εάν κάποιο κράτος έχει έλλειψη σε κτηνιάτρους, δεν είναι αυτό ο λόγος για να επιτρέπεται η έκδοση ε, συνταγής από έναν βοηθό κτηνιάντρου, κάποια άλλη λύση πρέπει να υπάρχει. Τα κράτη-μέλη λοιπόν που έχουν δυσκολία να εξασφαλίσουν επαρκή κάλυψη από κτηνιάτρους δεν πρέπει να επιτρέπεται να ε, δίνουν την άδεια σε ε, μη κτηνιάτρους να δίνουν συνταγές με την εξαίρεση των αντιπληκτικών. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Δεν ζήτησε άλλο κανεί το λόγο από του συναδέλφου. Έχουμε όμω τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση υγεία. Α, συγγνώμη πρώτα. Ε, ο κύριος Στράνκ είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλετε το λόγο, δεν είστε και υποχρεωμένος. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Trunk. Όχι trunk. το Για να απαντήσω στον κύριο Μπούντα. Σε σχέση με την ε, συνταγογράφηση φαρμακούχων ζωοτροφών. Η Επιτροπή προβλέπει τη δυνατότητα να μπορεί και κάποιος άλλος να συνταγογραφεί φαρμακούχες ζωοτροφές, αλλά αυτό με βάση το σύστημα που ισχύει στο κράτος μέλος. Θεωρήσαμε δηλαδή ότι είναι ζήτημα επικουρικότητας και ότι πρέπει το κάθε κράτος να εισακάγει ένα σύστημα που, όπως είπατε, έχει προβλέψει το Ρωμανό Βασίλειο. Εμείς υποστηρίζουμε μια τέτοια λύση. Και η διατύπωση που βλέπετε εδώ προκύπτει από τις συνομιλίες στο Συμβούλιο και, τη λιπές, και τις λοιπές ε, διαπραγματεύσεις με την κυρία Γκροστέτ. Για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Προτείνουμε λοιπόν να παραμείνει αυτή η επιλογή διαθέσιμη για τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τρόγκ. Οπότε ξαναδίνω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Γκιλέρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπε ο κύριος Μπούντα, που είναι σκιώδης συγητής για τον κανονισμό αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της προέβλεπε την ε, δυνατότητα συνταγογράφησης για τα ακτινατρικά φάρμακα, ε, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, στον τριμερή διάλογο, αυτή είναι η θέση που μας ε, παρουσίασε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον τριμερή διάλογο, η συμφωνία του Συμβουλίου είναι αρκετά περιοριστική σε ό,τι αφορά τα θέματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και όντως έγινε η συζήτηση, γιατί και στη Ρουμανία προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις ή κάποιοι επαγγελματίες που ε, έκαναν τις σχετικές ε, συνταγογραφήσεις. Το Συμβούλιο επισήμανε το πρόβλημα αυτής της κατάστασης. Και θα πρέπει να προσέξουμε ποιος δικαιούται να συνταγογραφήσει αντιβιωτικά ή κτηνιατρικά φάρμακα. Θα πρέπει όλα αυτά να είναι σωστά πλαισιωμένα και περιχαρακωμένα. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχει μια εξαίρεση λόγω της εθνικής νομοθεσίας που επέτρεπε αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό προβλέπει και η δική μας εντολή. Τώρα, μια ιδιαιτερότητα που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Ρουμανία ε, θα πρέπει να διευθετηθεί κάπως. Και εκεί έχουμε κάποιες διαφορές με το Συμβούλιο. Γιατί το Συμβούλιο ε, ζήτησε να έχει έκτακτο, εξαιρετικό χαρακτήρα λόγω της ιδιαιτερότητας του Ηνωμένου Βασιλείου και να ε, εξαλειφθεί σταδιακά. Πάντως, η εντολή που είχαμε ανέκαθεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένο αυτό το θέμα. Πάντως οι επαγγελματίες στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχαν τη δυνατότητα συνταγογράφησης προϊόντων, όχι αντιβιωτικών όμως, με σχετική πρόβλεψη της εθνικής νομοθεσίας. Αυτό καλύπτεται από την ιδιαιτερότητα, αλλά έχουμε μια εξαίρεση και στη Ρουμανία. Θα δούμε πώς θα το διευθετήσουμε το θέμα αυτό. Πάντως, ο εκπρόσωπος της Ρουμανικής κυβέρνησης ε, έπρεπε να είχε διεκδικήσει αυτό το θέμα πιο θερμά στο Συμβούλιο. Πάντως, όντως, προέκυψε ζήτημα. Θα δούμε τι λύση θα βρεθεί με τη Ρουμανία. Θέλουμε με βάση και την εντολή μας να καταλήξουμε σε σωστή λύση για να μην δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα. Και ε, η πρόβλεψη που είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο θα μας ε, χρησιμεύσει και στη συμφωνία με τη χώρα που θα έχουμε σε λίγους μήνες, αλλά και με τη Ρουμανία που είναι χώρα μέλος. Θα πρέπει να δούμε τι λύση θα βρούμε για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ωραία, δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε την κυρία Αγγιλέρα για την ενημέρωση έχουμε διεκπαιρεώσει σχετικά νωρίς το πρόγραμμά μας το πρωινό. Είναι 11 παρα 5. 11 και 4 θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τότε. Μέχρι τις 11 και 4. Παρακαλώ τους συνεργάτες να ενημερώσουν τους ε, συντονιστές ώστε να ξεκινήσουμε ένα τέταρτο νωρίτερα, δηλαδή σε 11 και 4 τη συνεδρίαση των συντονιστών. Και το απόγευμα πότε θα ξεκινήσουμε, τρεις, α όχι, όχι τρεις, συγγνώμη, δυόμιση η απογευματινή συνεδρίαση θα ξεκινήσει, δυόμιση το απόγευμα και 11 και 4 οι συντονιστές.